9 της σημερινή διάταξης. Θα το συζητήσουμε πριν από το σημείο 8. Το 9 λοιπόν θα το συζητήσουμε πριν από το 8. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν. Τι γλώσσες έχουμε σήμερα. Εσθονικά και μαλτέζικα δεν έχουμε. Όλες τις υπόλοιπες γλώσσες τις έχουμε. Δεύτερη ανακοίνωση στις 14 Μαρτίου μεταξύ 1 το μεσημέρι και 2.30 το μεσημέρι θα γίνει ένα εργαστήριο για την πρόληψη σε ό,τι αφορά θέματα υγείας. Και αυτό θα το παρουσιάσει ο κ. Πέτερ, λέει η κυρία Βίλμουτ. 4 Μαρτίου. Μεταξύ 1 το μεσημέρι και 2.30 το μεσημέρι. Ένα G2. Ύστερα, ε, τριμερή διάλογη στις ανακοινώσεις και πάλι, σε ό,τι αφορά την έκθεση Μακέβαν, το οποίο ολοκληρώθηκε ως θέμα στις 12 Φεβρουαρίου. ETS, έκθεση Πέτερ Λίζε, πρώτος τριμερής διάλογος στις 18 Φεβρουαρίου και μετά για την εξυγόνιξη της 18 Φεβρουαρίου έλαβε χώρα πρώτος τρομερής διάλογος και στις 4 Μαρτίου θα γίνει δεύτερη, ο δεύτερος τρομερής διάλογος. Μάλιστα, λοιπόν, να συνεχίσουμε. Έχουμε την οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Έχουμε το τροποποιημένο κείμενο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Περιβάλλοντος και σε ό,τι αφορά τις εξηγήσεις για τις αλλαγές. Το κείμενο λοιπόν αυτό θα το ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Και είναι λοιπόν αυτό ένα ολόκληρο πακέτο. Θα τα προσυπογράψουμε λοιπόν αυτά. Θα υπάρξει και μια επιστολή προς τον, προς τον ε, Πρόεδρο. Ωραία λοιπόν, αν δεν έχετε αντιρρήσεις έτσι θα προχωρήσουμε. Για τα πρακτικά τα οποία δεν τα εγκρίναμε. Τα πρακτικά λοιπόν της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2013. Δεν ξέρω αν υπάρχουν οποιασδήποτε αντιρρήσεις, ε, προσθήκες, όχι. Πολύ ε, ωραία. Πολύ Άρα λοιπόν εγκρίνονται έτσι τα πρακτικά. Και περνάμε λοιπόν στους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς. Μια ε, ψηφοφορία την οποία θα την διεξάγουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη λοιπόν της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εάν ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Τριντανέα ψήφι υπέρ. Εγκρίνεται λοιπόν. Και περνάμε τώρα λοιπόν στο σημείο 6 της ημερήσια διάταξης. Προφορική τροπολογία. Ξεκινάμε ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε για το κατά πόσο δεχόμαστε την ε, προφορική απάντηση. Δεν ξέρω αν ψηφίσατε όλοι. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται με τρεις ψήφους κατά. Ωραία λοιπόν. Και α περάσουμε τώρα στο σχέδιο ψηφίσματος. 13. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται πέπτη λοιπόν η επόμενη. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 17. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Παρακαλώ να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 17. ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Μάλιστα. Στην 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 34 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα να ψηφίσουμε από κοινού την 1 και τη 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά για τη 10. Έναρξη ψηφορίας. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να αλλάξουμε τη 12. Μάλιστα. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τη 12. Εάν ψήφισατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία παρακαλώ ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Και τώρα περνάμε έχουμε τη χαρά να ψηφίσουμε 1.200 τροπολογίες. Το συζητήσαμε και στους συντονιστές, το ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί. Η κυρία Χάση έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, μια λεπτομέρεια. Για την τροπολογία 1045 Εφόσον ε, έχει περάσει ενοποιημένη Επτά και από ό,τι είπε και ο εισηγητής δεν θα πρέπει να σημειώνεται ότι καταπίπτει μετά την ενοποιημένη 7. Έτσι είχαμε πει στις διαπραγματεύσεις με τους Σκιώδης. Μόνο στην τελευταία έκδοση του καταλόγου ψηφοφοριών σημειώνεται ότι καταπίπτει εφόσον περάσει η ενωπημένη ΣΕΒΑ και η ΕΠΤΑ, συγγνώμη, και θα θέλαμε αυτό να διορθωθεί. Να ψηφίσουμε την 1045 ως προσθήκη στην ενωπημένη ΕΠΤΑ. Ε, Έχω ενοχληθεί λίγο, λέει ο Πρόεδρος. Γιατί? Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε το κατάλογο ψηφοφορία λίγο πριν από την ψηφοφορία, αλλά να ρωτήσω τον εισηγητή αν συμφωνεί. Ε, ναι, εάν θέλουμε να την αλλάξουμε πρέπει να ψηφίσουμε για την πρόταση της συναδέλφου. Πρέπει να ψηφίσουμε επί της πρότασης. πριν γίνει η πρώτη ψηφοφορία. Σωστά. Σνέλχαρτ και μετά ο κ. Σνέλχαρτ. Ναι, να υποστηρίξω αυτό που λέτε, γιατί με την ενοποιημένη 7 δεν καλύπτεται η 1045. Άρα δεν καλύπτεται η τροπολογία αυτή από την ενοποιημένη τροπολογία αυτή. Είναι πάρα πολλές οι τροπολογίες στον αριθμό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήταν πάρα πολύ ε, σκόπιμο να την ψηφίσουμε την τροπολογία. Η κυρία Γκέρλινγκ. Thank you, Chair. Well, Θα θέλαμε να ψηφίσουμε την ενοποιημένη 8, παρακαλώ. Ναι, 18 μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν την ε, πρόταση αυτή και θα πρέπει να σηκωθούν. Δεν βλέπω να υποστηρίζεται αυτό το αίτημα. Εντάξει, θα δούμε αν φτάσουμε εκεί. Για την τροπολογία θα του χάσει ο κύριος Πυρίλο είπε να την ψηφίσουμε για την 1045 ως προσθήκη. Ποιοι είναι υπέρ αυτής της πρότασης. Κατά, παρακαλώ. Ηλεκτρονικά, άμα θέλετε. Άλλη μια φορά, παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης της Άτου Χάση για την τροπολογία 1045 προκειμένου να μην καταπέσει σε περίπτωση που η ενοποιημένη 7 εγκριθεί. Να ψηφιστεί ξεχωριστά. Όσοι είστε υπέρ της πρότασης της κυρίας Χάση, να ψηφίσετε το χέρι ψηλά. Ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά είναι πιο απλό, λέει ο πρόεδρο. Πιο απλό. τη πρόταση τη κυρία Σάτου Χάση. Ψηφίσατε όλοι. τη ψηφορία. Μάλιστα λοιπόν. Αυτό θα κάνουμε. Julie möchte über Consolidated Για την αναποιημένη 8 θέλει η κυρία Γκέρλιν να ψηφίσουμε ονομαστικά. Αν λοιπόν θέλει κάποιος να γίνει αυτό, θα πρέπει να σηκωθούν όρθιοι 18 συνάδελφοι. Κυρία Γκέρλινγκ. Μα σηκωθείτε, σηκωθείτε όρθια. Όρθια, όρθια, σηκωθείτε. Αν είσαστε αν υποστηρίζετε λοιπόν αυτή την πρόταση, ποιο είναι υπέρ να ψηφίσουμε ονομαστικά. Παρακαλώ να σηκωθείτε όρθιοι. Βλέπω ότι δεν σηκώνεται λοιπόν κανένα. Κυρία Γκέρλινγκ. Εάν θέλετε ονομαστική ψηφοφορία όπως και ζητήσατε, θα πρέπει να σηκωθείτε όρθια. Και εσείς και 18 συνάδελφοι στο σύνολο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τέσσερις συνάδελφοι. Τέσσερις συνάδελφοι λοιπόν. Πέντε. Δεκατρεις λιγότεροι από ό,τι χρειαζόμαστε. Δεν θα γίνει λοιπόν ονομαστική ψηφοφορία. Πολύ ωραία. Και τώρα ελπίζουμε, λέει ο πρόεδρος, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με τον κατάλογο ψηφοφορία. Να ξεκινήσουμε με την ενοποιημένη ένα. Ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Εάν ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. 36 υπέρ 8 κατά εγκρίνεται. Τροπολογή τροπολογία 125 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 140. Άγριο 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα συνεχίζουμε στο δεύτερο τμήμα. Στο δεύτερο τμήμα λοιπόν της 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα της 142 έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Άγκρι 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει. 143, 143 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 146 Έλεγχος, έλεγχος ζητείτε για το δεύτερο τμήμα της 145. Παρακαλώ, έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Στο δεύτερο τμήμα της 145. Αυτό ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 146 τώρα. Υπέρ παρακαλώ 146. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Okay. Dann müssen wir jetzt 106. Την 146 λοιπόν λέει ο Πρόεδρος τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 147, 148 καταπίπτουν το πρώτο τμήμα, αλλά το δεύτερο τμήμα πρέπει να ψηφιστεί. Υπέρ. Δεύτερο τμήμα λέει ο Πρόεδρος. 148 και η άγρια 9 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά για την 148 και την άγκρη 9 παρακαλώ ηλεκτρονική ψηφοφορία έναρξη πέρας απορρίπτεται 149 υπέρ κατά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 Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 167. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην ενοποιημένη 2. Ηλεκτρονικά επίσης. Έναρξη. Πέρας. εγκρίνεται με σαφή διαφορά. Και συνεχίζουμε λοιπόν τώρα. Με την 177. Συνεχίζουμε. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 178 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται το 11 Α, ήταν η ίδια, ήταν η ίδια, ταυτόσημη. Πολύ ωραία. 179 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άκρη 12, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 180, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 181, υπέρ. Έλεγχος για την 180. Ωραία. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 180. Πέρας. Απορρίπτεται. 181, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 182 ναι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 185 και άγκρι 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 186 και άγκρι 14 υπέρ. Κατά. Απόχες. Να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. 186 και άγκρι 14 παρακαλώ. Ένα ψηφοφορίας. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα συνεχίζουμε με την 187 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 188 και άγκρι 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 189, άκρη 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. άκρη 18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 191 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 192 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 196-197 ε, συμβατές. Από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 198 καταπίπτια. Άγκρι 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 199 και 200. Υπέρ. Α, και 201 μαζί. Και 202. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τις τέσσερις μαζί παρακαλώ να τις ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. 199 μέχρι 202. Είναι γλωσσοϊκό το θέμα. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 203. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 204, 205, 206. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφέ το αποτέλεσμα. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 204 έως 206. Παρακαλώ ηλεκτρονικά. Έναξη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 207 και άκρη 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 208 άγκρι 21. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 211 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 212 υπέρ. Κατά. Αποχές τα 213 υπέρ. Κατά. Αποχές. Κουραστήκατε. Κουραστήκατε. Έχουμε ακόμα 92 σελίδες. Ηλεκτρονικά. Για να το ελέγξουμε παρακαλώ. Και τη 213. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 214. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρη 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 215. Καταπίπτει. Α, 215. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 216 και άγκρι 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συνολικά να κοιτάξουμε τη 217, 218, 219 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 220 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 221 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 222 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 223 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 224. Έχουμε ψηφοφορία σε τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Χωρίς Μάλλον πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα το σύνολο του κειμένου και μετά τη λέξη single. Πρώτα λοιπόν το σύνολο του κειμένου. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και έτσι το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Άγκρι 24. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 25 άγκρι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 225. Υπέρ. Α, καταπίπτει. Η 226. Ψηφίζουμε την 226 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και τώρα συνεχίζουμε την 231. Άγκρι 27, 232, 233. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 234. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα συνεχίζουμε με την ενοποιημένη 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 251 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 252 υπέρ. Α, και 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 253 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 254, 255 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ενοποιημένη. Α, να ελέγξουμε την 255, λέει ο Πρόεδρος. Την 254 και την 255. Ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφορίας, αν ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Ενοποιημένη 4, ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Έναρξη ψηφορίας. Για να ψηφίσατε όλοι. Πέρα ψηφορίας. εγκρίνεται. Και τώρα λοιπόν περνάμε στη σελίδα 17, σε στο δικό μου κείμενο, τροπολογία 281-293. Αυτές οι δύο. 281-293, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 282, άγκρι 36, υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. 282 και 36. Έναρξη. Πέρασε. ...283 απορρίπτηκε. 283 άγκρι 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 284 υπέρ Κατά. Αποχές έγκρινεται. 285. Άγκρι 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και συνεχίζουμε με την... Με την 289. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 290. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 291 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 292 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 294 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 295 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 296 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 297 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 298 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 299 υπέρ. Α, καταπίπτει. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Α, όχι, δεν ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε. Την 299 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 300 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 301 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 302 καταπίπτει. Η 303 επίσης. Άγκρι 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 304 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 305 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται η 306 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 300 να ελέγξουμε την 307 να ψηφίσουμε παρακαλώ υπέρ Κατά. Άποχες απορρίπτεται 308 υπέρ. Κατά. Άποχες έγκρινεται 309 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Άγκρι 40. Σε δύο τμήματα παρακαλώ. Α, δεν ψηφίζεται το δεύτερο τμήμα, το δεύτερο τμήμα της Άγκρη 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 310. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 311. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 312. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3.15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 3.17 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 41, πρώτο τμήμα. Δεν ψηφίζεται. Άγκρι 41, δεύτερο τμήμα λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 318, υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 318 έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισατε όλοι. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 319 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 320 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 321 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 322. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 323. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 324. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μπλοκ 4 υπέρ, κατά, άποχες. Ξανά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ για το μπλοκ 4. Haben alle abgestimmt? Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Ενοποιημένη 5 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε με την ενοποιημένη 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 3.48. Δεν ψηφίζουμε για την 3.48. Άγκρι 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Παρακαλώ την Άγκρη 45 να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μεγάλη διαφορά. Άγκρη 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρη 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 360 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται 361 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 362 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 363 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 364 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 365 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 366 367 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άκρη 48 πρώτο τμήμα υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 368 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 369 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 370 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 371 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 372. Άγκρι 49. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 373. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 374 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 375 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε παρακαλώ τον 375 ηλεκτρονικά. Ένα ηλεκτρονικής ψηφορία Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. η 376 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 377 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 378 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Η 379 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Μπλοκ. 5 υπέρ. Κατά. Κατά, απορρίπτεται. Τρία δύο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 384 και άγκρι 50. Υπέρ. αποχές απορρίπτεται. Η 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 386 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 387 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 388 ναι, την ψηφίζουμε. Α, καταπίπτει. Καταπίπτει. Η 20 παρακαλώ. Να ψηφίσουμε την 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 389. Και η άκρη 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 390 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 391 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 392 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 393, 394, 395, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εναποιημένη 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε στη σελίδα 34. Κυρία Στέχαρτ, ο κύριος Σνέχαρτ, συγγνώμη. Έχουμε ε, λοιπόν ε, την απόφαση που πήραμε προηγουμένως να ψηφίσουμε ως προσθήκη την 1045, θυμάστε? Ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Αλλά έχουμε φτάσει στην 442 στη σελίδα 34, παρακαλώ. Υπέρ.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 Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 446. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 447 υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Και τώρα να ψηφίσουμε την 448 και την άκρη 53 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 449. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 450 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 453 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 452 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 454 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 455 Άγκρι 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 456 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 457, 458. Ταυτόση μέσα από κοινού λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 459, 460, Άκρη 55 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 461 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, το Συμβούλιο. Το εγκρίνεται. 462 Άγρι 56 περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 463. Σε δύο τμήματα παρακαλώ. Πρώτο τμήμα. Καταπίπτει. 464 υπέρ. Δεύτερο τμήμα ως προσθήκη. 463, δεύτερο τμήμα, διορθώνει πρόεδρο. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχέ έγκρινεται. 464. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 465. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 466. Υπέρ. Κατά. Αποχέ έγκρινεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 467 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 468 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 469 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 470 471-472. Από κοινού τις ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, γι' αυτό λοιπόν να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 473. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 474. Άγκρι 57. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 474 και την άγκρι 57 ηλεκτρονικά. Έναρξη. Αν ψηφίσετε όλοι, πέρασε. Απορρίπτεται. Το επόμενο άρθρο το ψηφίζουμε. Περνάμε λοιπόν στην 478. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Να το ελέγξουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε με την τροπολογία 480. 480 παρακαλώ ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 481 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πρόβλημα υπάρχει σε ό,τι αφορά τα αγγλικά. Vielleicht darf Να μιλήσω, να μιλήσω, συνάδελφε. Πρόβλημα με την αγγλική μετάφραση. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την ισπανική διερμηνία. Δεν δουλεύει η ισπανική καμπίνα. Είναι 481. Εντάξει, όλα καλά λέει ο πρόεδρος. Όλα καλά. «481 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 482 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 483 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 485 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 484 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ηλεκτρονικά την 484 παρακαλώ. Εάν ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 486 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 487 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 488 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 489 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν είναι σαφές. Παρακαλώ, ας το ελέγξουμε. Γιατί είναι 489. Παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 490. Μπλοκ 6. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 492. Ε, Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 493. 494. Τι έγινε με τι μηχανε 493 493-494 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 495-496 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 58 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 497 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 498 και άγκρι 59 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 506 παρακαλώ. Μπλοκ 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 501 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν είναι σαφές. Παρακαλώ να ελέγξουμε την 501. Έναρξη ψηφοφορίας. Αν ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 503 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 504. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 505. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 506. Ein Προφορική τροπολογία από το ΕΛΚ. Αυτό ψηφίζουμε λοιπόν τώρα. Κύριε Να εξηγήστε μας. Ναι, κοιτάξτε, στο άρθρο 23, στο σημείο 4, θεωρώ ότι πρόκειται για μια γενική εξουσιοδότηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναφέρεται ότι οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση μπορούν να αποκλίνουν από όλα όσα έχουν αποφασιστεί έως τώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό θεωρώ, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω να υποστηρίξετε τη διαγραφή του κειμένου αυτό, σε ό,τι αφορά δηλαδή την έγκριση της τροπολογίας 507. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Να το ψηφίσουμε. Πρόφορο και τροπολογία 507 υπέρ. Κατά. Με μεγάλη πλειοψηφία υποστηρίζεται λοιπόν, εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 509. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 510. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 511. Άγκρι 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές απο, ε, ναι. Προφορική τροπολογία 1. Στην 512. Υπέρ. Κατά. Μόνο οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι συμμετείχαν σε αυτή την ψηφοφορία. Σας παρακαλώ πάλι πάμε. Παρακαλώ ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Για την προφορική τροπολογία 1 στην τροπολογία 512. Έναξη ψηφοφορίας. Ψηφίσετε όλοι. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 20 είναι υπέρ, 8 κατά. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με την 512. 514 ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 515. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Έγκρινεται. Η 516. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 517. Καταπίπτει. 518. Υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 519 καταπίπτει, 61, άγκρι 16 καταπίπτει και 520. Άγκρι 62. Τραπολογία 521, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 522, ε, υπέρ. Α, όχι. Η 522. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 523, 524, ε, 63 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 525 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 526 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 527. Καταπληκτή. Και αυτή. Η 528. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 529, τα 65 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 531 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η τροπολογία. Η 530 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 532 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 533 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 534 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 536 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 537 άγκρι 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μπλοκ 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 541 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 542 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 543 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται 544, αύριο 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 545 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι καλύτερα να την ελέγξουμε παρακάτω την 545 ηλεκτρονικά. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η 31 υπέρ. Εγκρίνεται. 546 υπέρ. Α, καταπίπτει. 547 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 548 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ή 549 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Παρακαλώ να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 549. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Με σαφήνεια. 550. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 551. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 552 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 553 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Άκρη 69 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 32. Κατά Καταπίπτει. 554 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπέρ 555 το δεύτερο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 556, 557 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 558 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Άκρη 70, συγγνώμη, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άκρη 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άκρη 72 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άκρη 73 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 559 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 74. Μπλοκ 9. Συγγνώμη. Μπλοκ 9. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Παρακαλώ ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τον μπλοκ 9. Εάν ψήφισατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 560 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 561 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Να ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 561. Εάν ψηφίσατε όλοι, Πέραστη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 562, άγκρι 76, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 563 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 564 αγκρίβονται 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 565 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Η 567 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι. Άγκρι 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 568 και άγκρι 79 υπέρ. Κατά αποχές απορριφθήκε. 569 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 570 Α, καλύφθηκε, εκπίπτει. 81, υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίφθηκε. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν μετά από έτοιμα Σνέρχαρτ, Άγκρι 81 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Πράγματι εγκρίθηκε. Άγκριο 82. Για να είμαστε βέβαιοι θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Σε δύο τμήματα. Σε δύο τμήματα. Την 571 σε δύο τμήματα. Υπέρ. 571 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 572 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 573 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 574 δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε 575 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 576 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 577 στο δεύτερο τμήμα υπέρ το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Απόχες. Δεν είναι σαφές. 577 δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγ... Απορρίφθηκε λέει ο Πρόεδρος ισοψηφία. Μπλοκ 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα τις 579 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 580 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 582 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 583 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 584 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 585 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 586 έως 589 υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν καταπίπτει 590 ή 591 δεύτερο τμήμα και τρίτο τμήμα πρέπει να ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 591 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Τρίτο τμήμα. Θα ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα. Εντάξει. 591 δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Ισοψηφία. Τρίτο τμήμα της 591 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 593 δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε. Η 33 τροπολογία υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίθηκε. Άγκρι. Α, η 83 καταπίπτει. Εντάξει, 34 και άγκρι 84 υπέρ αυτών κατά άποχες εγκρίθηκαν 500 Είχε εγκριθεί η άλλη. Α, δεν χρειάζεται να ψηφιστεί αυτή. Εντάξει. Η 595 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 596 άγριο 86 υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν 597 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 598 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Λοιπόν, κάναμε τα μισά περίπου και έχουμε μια ώρα, μια μισή ώρα σχεδόν σε ψηφοφορίες. Πρέπει να συζητήσουμε πώς εργαζόμαστε όσον αφορά πίνακες καταλόγους ψηφοφορίας, χρόνο ψηφοφορίας και όλα τα λοιπά. Το παρακάνουμε. 599, δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 600 δεύτερο, ε, πρώτο τμήμα υπέρ 600 πρώτο τμήμα δεύτερο τμήμα της 600 δεύτερο τμήμα της 600 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 602 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 603 και άγριο 87 υπέρ αυτών κατά αποχές δεν είναι σαφές 603 και άγριο 87 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκαν η 604 τώρα. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 605 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 606 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Μπλοκ 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 610 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 36 λοιπόν ελέγχουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Η 611 και άγριο 88 υπέρ αυτών. Κατά. Αποχές. Ασαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε 611 και άγριο 88 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα α, απορρίφθηκαν. Η 612 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Μπλοκ 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 617 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 620 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές 620 λοιπόν ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα απορρίφθηκε η 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 619 υπέρ κατά άποχες απορρίφθηκε. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 619 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε. Μάλιστα. Η 621 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε μπλοκ 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε μπλοκ 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Άγκρι 627. 627 υπέρ. Κατά. 628 λοιπόν. 628 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 629 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Μπλοκ 15 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 634 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 635 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 636 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 637 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 638 σε τρία τμήματα το δεύτερο τμήμα θα ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 639 δεν θα ψηφιστεί συνεχίζουμε 640 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 642 και άγρια 96 υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν 600... να ελέγξουμε εντάξει 642 και άγρια 96 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκαν μάλιστα εγκρίθηκαν 643 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 644 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 645 άγκρι 97 υπέρ αυτών. Κατά αποχές απορρίφθηκαν. 646 άγκρι 98 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκαν. 647 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 648 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 649 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 650 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 651 άγρια 99 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν άγρια 100 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ψηφίζουμε την άγρια 100 ηλεκτρονικά άρχεται άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα εγκρίθηκε πάμε στην μπλοκ 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 654 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 657 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 658 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Άγκρι 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 659 και 660 δεν είναι ταυτόσιμες. Πρέπει ξεχωριστά να ψηφιστούν οι κάθε μια. Η 659 πρώτα υπέρ κατά αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε την 659 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 660 τώρα και η 661 υπέρ κατά θα ελέγξουμε 660-661 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία επ' ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκαν 662 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 662 λοιπόν θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία επ' αυτής. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Ισοψηφία απορρίφθηκε. Πάμε στη συνέχεια στην 663 και 664 υπέρ αυτών. Κατά αποχές απορρίφθηκαν. 665 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 666 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 667 ξεχωριστά η 667 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 668 και 669 από κοινού υπέρ κατά αποχές. Ασαφές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. 668, 669. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκαν. Οι 670 και άγριοι 102 υπέρ αυτών. Κατά αποχές εγκρίθηκαν. 671 υπέρ. 671 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 672 και 673 υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν θα ελέγξουμε εντάξει 672-673 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας Απορρίφθηκαν. Μάλιστα. 674 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 675 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 676 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 677 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 677 ηλεκτρονικά άρχεται εντάξει άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας και απορρίφθηκε μάλιστα 678 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 679 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 680 υπέρ κατά απορρίφθηκε 681 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 682 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 683 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 684 και άγρια 103 υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν 685 και άγρια 104 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 686 και άγρι 105 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. Μπλοκ 17 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Μπλοκ 18 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 693, 94 και 95 από κοινού οι τρεις υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκαν. Να ελέγξουμε. Εντάξει, ψηφίζουμε 693, 94 και 95 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκαν, μάλιστα, εγκρίθηκαν. Πολύ καλά. 696 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Συνεχίζουμε με την εντεταγμένη 8 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. «714 τώρα. Α, δεν θα, θα ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Και πάλι ψηφίζουμε στη σελίδα 61 στον κατάλογο μου εδώ στον πίνακά μου την τροπολογία 714. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 714 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 64-39 υπέρ. Στη σελίδα 64, σελίδα 64, η 39 τροπολογία. Σελίδα 64, τροπολογία 39. Στη δική μου σελίδα είναι η σελίδα 64 στον καταλογό μου. Τροπολογία 39. Υπέρ λοιπόν. Υπέρ της 39. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Άγκρι 112 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Άγκρι 113 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές 113 άγκρι ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι Πέρας ψηφοφορίας και απορρίφθηκε. Θα κάνουμε ένα άλμα τώρα. Σε μένα είναι η σελίδα 72 στον κατάλογό μου. Σελίδα 72. Τροπολογία 805, 806, 807 και 808 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν Με 100 τόσες σελίδες μπορεί κανείς να χάσει τον μπούσουλα. Συνεχίζουμε με την τροπολογία. Agri 119. 119. Agri 119 τροπολογία που πρέπει να ψηφίσουμε. Άγκρι 119. Η 76, σελίδα 76 στον καταλογό μου. Άγκρι 119 τροπολογία. Άγκρι 119. Τα βρήκατε, την βρήκατε την τροπολογία αυτή, υπέρ λοιπόν κατά αποχές εγκρίθηκε 120 άγριε 120 υπέρ α όχι 851 λοιπόν τροπολογία υπέρ κατά αποχές ασαφές το αποτέλεσμα ψηφίζουμε την 851 ηλεκτρονικά άρχεται Λοιπόν, πολύ καλά. Τι γίνεται με το, τη συσκευή εκεί. Πολύ καλά. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. 19 υπέρ 20 εναντίον απορρίφθηκε λοιπόν. Και αλλάζουμε προεδρία. Παρακαλώ. Τα υπόλοιπα να τα ψηφίσουμε ομού όλα για να τελειώνουμε, μια και έξω. Ε, λοιπόν, 851 τροπολογία τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Να ελέγξουμε. Η ψηφοφορία άρχεται. 851. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Μάλιστα. Απορρίφθηκε. Πολύ ωραία πρώτη ψηφοφορία για μένα ως αποτέλεσμα. 852 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. 853 ε, ψηφίζουμε υπέρ. Κατά από, εγκρίθηκε 854 και άγκρι 121 από κοινού υπέρ αυτών κατά αποχές θα ελέγξουμε 854-121 ηλεκτρονικά άρχεται πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκαν 855 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Άγρι 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Άγρι 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 856 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 857 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 800 να ελέγξουμε 857 άρχεται ηλεκτρονικά 857 πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε η 857. Λυπούμε, καθυστερήσατε πολύ. Υπήρχε επαρκής χρόνος για να ψηφίσετε, να συμμετάσχετε. 858 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 859 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 860 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε να ελέγξουμε 860 άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε μάλιστα εγκρίθηκε τροπολογία 862 και άγρια 124 είναι ταυτόσιμες υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 863 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 864 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 865 και άκρη 125 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν τροπολογία 44 υπέρ αποχές εγκρίθηκε 866 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 867 και άγρια 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν 868 και άγκρι 127 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 869 και 870 υπέρ αυτών κατά αποχές θα ελέγξουμε 869-870 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκαν πράγματι, εγκρίθηκαν. 871 και 872 υπέρ αυτών. Κατά αποχές Να ελέγξουμε και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία 871-872 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Και εγκρίθηκαν πράγματι. Τροπολογία 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 873 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ασαφές το αποτέλεσμα και πάλι. Ελέγχουμε. 873 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας πληφοφορίας. Εγκρίθηκε αυτή. Εντάξει. Οι επόμενε δύο ομάδες ε, έχουν εγκριθεί οι τροπολογίε του. Πάμε στην 880 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίφθηκε. 881 και άγρια 128 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 882 και 883 και block vote υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν 884 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 885 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 886 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 887 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 888 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 889 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 890 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 891 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 892 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 893 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 47 και 48 block vote υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν. 894 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 895 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 896 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 897 και 898 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 899 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 900 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 901 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε μπλοκ 23 902 δηλαδή και 903 και 904 τροπολογίες υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν 905 τώρα υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε. Τροπολογία 50 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε. 906 υπέρ κατά απόχες να ελέγξουμε. 906 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας, εφόσον ψηφίσατε όλοι, και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Η 907 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 908 και άγκρι 129 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. 909 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 910 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 910. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέ, πέρας ψηφοφορίας τώρα. Εγκρίθηκε αυτή η τροπολογία. Η 911 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και πάλι θα ήθελα να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 911. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίθηκε η 911. Μάλιστα. Η 912 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίφθηκε. Η 913 και άγρια 130 υπέρ αυτών. Κατά. Απόχες. Εγκρίθηκαν. Η 914 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίθηκε. Να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 914 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 915. 915 και 916 ομού υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκαν 917 υπέρ να ελέγξουμε εντάξει ψηφίζουμε την 916 προς έλεγχο άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 915-916 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα απορρίφθηκαν πράγματι. Τροπολογία 917 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίθηκε. 918, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίθηκε. 919, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίφθηκε. 920, υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε ε, να ελέγξουμε ελέγχουμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 920 άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας και απορρίφθηκε πράγματι Προπολογία 921 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 922 και 923 υπέρ αυτών κατά αποχές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά προς έλεγχο 922-923 άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα απορρίφθηκαν Η 924 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε μπλοκ επί της 925 μέχρι κάτω την 948 υπέρ αυτών όλων κατά αποχές απορρίφθηκαν η 926 και η άγρια 131 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. Η τροπολογία 929 και η άγρια 132 υπέρ αυτών. Κατά αποχές απορρίφθηκαν. Η 930 και άγρια 133 υπέρ αυτών. Κατά αποχές εγκρίθηκαν. Η 933 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 935. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Ζητήσατε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 935. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και εγκρίθηκε το δεύτερο τμήμα της 935. Μάλιστα. Και τώρα θα πάμε στην 938 και άγκρι 134 υπέρ αυτών. Κατά οι σοσιαλδημοκράτες. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, αφού οι σοσιαλδημοκράτες ε, αποφάσισαν πως θέλουν να ψηφίσουν τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία, 938-134 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Εγκρίθηκαν. Μπλοκ 25, 939 μέχρι 935-936 άγκρι. Υπέρ αυτών. Κατά. Απορρίφθηκαν. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Μπλοκ 25. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκαν πράγματι. 940 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Η 941 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Η 942. Έλεγχος λέτε. 941. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε λοιπόν. Εγκρίθηκε. Τώρα η 942 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 944 και άγκρι 137 υπέρ αυτών κατά αποχές έλεγχος ψηφίζουμε 944 και 137 άγκρι άρχεται Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας και απορρίφθηκαν σαφώς. Τροπολογία 947 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Η 949 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Η 950 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε την 950 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Και εγκρίθηκε. Η 951 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 952 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 953 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 954 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 955 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 956 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 957 και άγκρι 138 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 958 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε την 958 ηλεκτρονικά προς έλεγχο. Άρχεται. Λυπούμε. 959 εντάξει. Α, όχι. Είχα δίκιο. Είχα δίκιο. 958. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 958. Σωστά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίθηκε. Η 139 καταπίπτει, πίπτη, 139. 959 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 960, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 961, υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε 962 και 963 ταυτόσιμες υπέρ αυτών κατά αποχές ελέγχουμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά 962-963 άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκαν αυτές η 964 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 965 και 966 υπέρ αυτών. Κατά αποχές απορρίφθηκαν. 967 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 968, 969 και 970 υπέρ αυτών. Κατά αποχές απορρίφθηκαν. 971 Έλεγχος. Ψηφίζουμε την 968, 969, 970. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορία τώρα. Απορρίφθηκαν. Η 971, 972, 973. Υπέρ αυτών. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκαν. 974 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 975 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε μπλοκ 26 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε μπλοκ 26 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκαν η 983 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Μπλοκ 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποχές. Συγγνώμη. Απορρίφθηκε. 989 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ασαφές το αποτέλεσμα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Την 989. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 990 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 991. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε αυτό πίστευα κι εγώ. Εντάξει, να ελέγξουμε. Δεύτερο τμήμα τη 991. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Και απορρίφθηκε πράγματι. Δεν θα ψηφίσουμε την άλλη. Η 993 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 995-996, μπλοκ 28. Υπέρ αυτών. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκαν. Τροπολογία 997. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 997 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε λοιπόν το δεύτερο τμήμα. Το τρίτο τμήμα της 997 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίφθηκε, αλλά θα ελέγξουμε το τρίτο τμήμα ηλεκτρονικά της 997. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε, εγκρίθηκε με την ίδια πλειοψηφία. Τροπολογία 999 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 1000 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 1001 υπέρ κατά αποχές, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε μπλοκ 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1004 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1005 συμβατή. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1006 και άγκρι 142. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1006 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1009 και 1011 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 1009-1011 άρχεται η ψηφοφορία εψήφισαν άπαντες πέρας απορρίπτονται 1008 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 1010. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1000. Ελέγχουμε για τη 1010. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 1012. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1013 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1014 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1015 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1016 και 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1018 και άγκρι 143 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1019 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1020 και 1025 καθώς και άγκρι 145 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1021 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1022 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1023 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1024 υπέρ, έλεγχος για την 1023, άρχεται η προφορία. Εψήφισαν άπαντες, πέρας. Απορρίπτεται. 1024 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1026 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1027 και 1028 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1029 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1030 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1031 υπέρ κατά αποχές Απορρίβεται. Έλεγχο. Θέλετε έλεγχο. Θέλετε κύριε Σνέλχαρτ. Εντάξει. Θα το θυμηθώ την επόμενη φορά που το ζητήσετε. 1032 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 1034. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίβεται. 1033 πρώτο, δεύτερο μάλλον και τρίτο τμήμα. Όχι. Ξεκινούμε με το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εντάξει, να κάνουμε έλεγχο για το δεύτερο τμήμα της 1033. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα της 1033 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1037 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1040 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1041 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 1042 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1043 και άγκρι 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε για το 1043 άγκρι 149 Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Απορρίπτεται. 1044. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε την 1045. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1047 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε γιατί το ΕΛΚ ψήφισε διαφορετικά αυτή τη φορά 1047 άρχεται η προφορία πέρας εγκρίνεται. 1046 και άγκρι 150 καταπίπτουν. 1048 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1049 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1050 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 1051 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1052 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1053 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1054 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1055 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 1056-1057 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τις 1058, 1059 και 1060 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Καλά λοιπόν, ας ελέγξουμε 1058, 59 και 60. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1061 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1062 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1063 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1064 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1065 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Φτάνουμε στα παραρτήματα. 1066 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1000 Ελέγχουμε το 1066. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνονται. Ευχαριστώ το ΕΛΚ για την προσφορά του. Ψηφίζουμε την 1067 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 68, στο τέλος της συνέδεσης 95 της δικής μου, του δικού μου καταλόγου ψηφοφοριών υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 70 υπέρ. Η 69 καταπίπτει. 70 και πάλι υπέρ. Βάσει της γραμματείας το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Περνάμε στην 70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 71. Μόνο το τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά να ελέγξουμε για το τρίτο τμήμα της 71. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Απορρίπτεται. 72. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε για την 83. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε για τον 85. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 88 και άγκρι 2. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 95 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε για την 95. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Ψηφίζουμε για την 97 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 99 και άγκρι 3 υπέρ. Κατά αποχές. Να ελέγξουμε για την 99 άγκρι 3. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 100 υπέρ κατά αποχές αγκρίνεται. Πρώτο τμήμα της 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα της 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πρώτο τμήμα της 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε για την 110 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες πέρας και εγκρίθηκε με 29 προς 6 και μία αποχή. Έχουμε και την τελική ψηφοφορία για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε με 25 προς 5. Συγχαρητήρια Συγχαρητήρια στον συγκεκριτή. Okay, we, we lost a lot of time. Χάσαμε πολύ χρόνο με τις ψηφοφορίες, οπότε παρακαλώ να φύγετε από την αίθουσα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, εάν δεν σας ενδιαφέρουν το σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή η χωστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων. Ο Στρέν Στίβενσον θα μιλήσει εκ μέρους του κυρίου σκι, οπότε να το δώσω το λόγο αμέσως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Ριτσχή στέλνει τις, τη δήλωσή του, διότι δεν μπορούσε ο ίδιος να έρθει. Η παρούσα πρόταση έχει συμφωνηθεί μεταξύ των θεσμικών οργάνων και ε, των κατομελών του 2013 μετά την έγκριση της ε, θέσης του Κοινοβουλίου με πρώτη ανάγνωση το 2013 και με τροπολογίες που προέκυψαν μετά από τις διαπραγματεύσεις του Μερούς Διαλόγου το Σεπτέμβριο του 2013. Παρόλο που το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων εγκρίθηκε από αυτή την Επιτροπή το Νοέμβριο του 2013 και με ευρεία πλειοψηφία, 45 ψήφους υπέρ και μόνο 11 κατά, είναι απαραίτητο, πρωτού περάσουμε στη δεύτερη ανάγνωση και την ολομέλεια, να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολή τροπολογιών σε επίπεδο επιτροπή. Ενώ ε, σεβόμαστε πλήρω τι διαδικαστικέ αυτέ ε, περιπλοκότητε ε, και ενώ σεβόμαστε το δικαίωμα κάθε βουλευτό να υποβάλει τι τροπολογίε του για να επιδιώξει του δικού του πολιτικού στόχου, ω υπεύθυνο εισηγητή για το φάκελο, για το θέμα αυτό, σα ζητώ να μην το κάνετε μέχρι την άνοιξη των επίσημων διαπραγματεύσεων. Ε, ο λόγος είναι τρίπτυχος. Πρώτον, οποιαδήποτε αλλαγή θα ε, καταστρέψει τη συμφωνία μας και θα εκθέσει εμάς, το μελλοντικό κοινοβούλιο καλύτερα, θα, θα μας φέρει σε μακροσκελείς διαπραγματεύσεις, ενώ είναι απαραίτητος και άμεση η ανάγκη επικαιροποίησης αυτού του κανονισμού και μάλιστα δεν βρισκόμαστε στο ύψος των διεθνών προτύπων αυτή τη στιγμή. Ε, κατά δεύτερον, ως ε, εισηγητής, συνείδησα ένα ε, ασυνήθιστα ενωμένο στις απόψεις του Συμβούλιο, το ίδιο και την Επιτροπή να συμπαρατάσσεται μαζί τους. Οι αλλαγές στο τωρινό κείμενο ήταν ε, κάποιες αλλά περιορισμένες. Και τρίτον, το συμπεφωνημένο κείμενο αξίζει να υποστηριχθεί, ακόμη και αν η θέση του Κοινοβουλίου ήταν φιλοδοξότερη από κάποιες ε, σκοπιές. Για να δώσω ορισμένα παραδείγματα, συμφωνήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, εκπονεί μελέτης αντικτύπου για τα θέματα της επισήμανσης και για τον τομέα της ηχορύπανσης με σοβαρές πληροφορίες. Οι κατασκευαστές υποχρεώνται να παράσχουν πληροφορίες για την ηχοστάθμη στα οχήματα, στο σημείο πώλησης και με τις τεχνικές ε, προδιαγραφές που πρέπει να διαπούν τα υλικά τους. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για την κατάταξη της δυνατότητας οδήγησης και ε, για την ηχοστάθμη βάσει των στοιχείων που τις παρέχουν τα κράτη-μέλη. Κάτι που ήταν ούτως ή άλλως πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο. Ένα σύστημα προειδοποίησης για τα ευρυδικά και τα ηλεκτροκίνητα οχήματα θα γίνει υποχρεωτικό μέσα σε μια τριετία βάση και μετά από τη θέση σε ισχύ του κανονισμού και σε πέντε χρόνια για όλα τα οχήματα αυτού του τύπου. με την ε, κίνηση της μηχανής θα ισχύει το σύστημα αυτό στην ουσία και αυτό θα έπρεπε να ικανοποιεί το Κοινοβούλιο. Επίση, οι οριακές τιμές που καταφέραμε να επιτύχουμε φτάνουν τα 68 δεσιμπέλ για τα πλέον συνηθισμένα επιβρατικά οχήματα ε, και φαίνεται να είναι φιλόδοξο αλλά από, είναι από τεχνικής πλευράς είναι εφικτός στόχος και βιώσιμος. Πολλοί από από εσά μπορεί να βρήκατε το στόχο αυτό όχι αρκετά φιλόδοξο. Να σα θυμίσω την μελέτη τη TNO, ενό ανεξάρτητου ιδρύματο, που βρήκε ότι οι οριακέ τιμέ που εγκρίθηκαν κατά τι διαπραγματεύσει, συγκρινόμενε με την τωρινή κατάσταση, είναι πολύ σημαντικέ για τι πέντε βασικέ κατηγορίε οχημάτων. 2,8 ε, δεσιμπέλ χαμηλότερα είναι οι σημερινές τιμές. Όμως το Φεβρουάριο του 2013 αυτό το που πρότεινε το Κοινοβούλιο ε, ε, είναι χαμηλότερο μόνο κατά 1,9%. Η διαπραγματευτική διαδικασία ήταν δυσκερή, Όμω νομίζω η τελική συμφωνία θα πρέπει να είναι ικανοποιητική για όλου. Ε, για όλου του άνωθοι λόγου, λοιπόν θα έλεγα να στηρίξουμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εμεί ευχαριστούμε κύριε Στίβενσον. Μα τελειώνει ο χρόνο. Η πρότασή μου είναι να δώσουμε ένα λεπτό στους κοιόδης στην κατάλογο μου έχω τον κύριο Ταταρέλα και τον κύριο Κράμερ και την κυρία Μέρκης. Κύριε Ταταρέλα. Και λιγότερο, αν θέλετε, Πρόεδρε, γιατί το συζητάμε τρία χρόνια το θέμα αυτό. Νομίζω ότι το θέμα έχει οριμάσει πλέον και ο στόχος δεν είναι να μπούμε πλέον στο περιεχόμενο, αλλά να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να περάσει ο κανονισμός αυτός ή όχι διότι εμείς είμαστε υπέρ του να εγκριθεί. Οπότε θα έλεγα οι συνάδελφοι να απόσχουν από περαιτέρω τροπολογίες. Ευχαριστούμε κυρία Μέρκης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ειλικρινώς πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα δυστυχώς διότι ο θόρυβος είναι ένα υποτιμημένο πρόβλημα και η χορύπανση έχει συνέπειες και στην υγεία, ιδίω σε, περιοχές, σε ανθρώπους που ζουν σε μειονεκτούσες περιοχές. ιδίω σε δρόμους με πολλή κίνηση και με οικογένειες χαμελού εισοδήματο. Γι' αυτό θα έπρεπε να επιδιώξουμε μια φιλόδοξη και ρεαλιστική στρατηγική για να μειώσουμε το επίπεδο ηχοστάθμιση των οχημάτων, για να προστατεύσουμε και τι κοινωνικέ μα αξίε αλλά και την ανταγωνιστικότητα τη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη. Αυτό δεν συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία θα μπορούσαμε να είχαμε υπάρξει πολύ περισσότερο φιλόδοξη και ήταν πιο φιλόδοξη από το Κοινοβούλιο η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα, ε, στοιχεία, υπόψη όλα τα στοιχεία της επιτευχής της συμφωνίας, η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη από την τωρινή, γι' αυτό και θα αναγκαστούμε να δεχτούμε το τελικό αποτέλεσμα, την συμφωνία αυτή. Όμως εμείς προτείναμε φιλοδοξότερη προσέγγιση για τις οριακές τιμές Πιστεύουμε ότι και το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να είναι καλύτερο και οι οριακές αξίες θα μπορούσαν να ήταν φιλοδοξότερες. Μια, ένα παράδειγμα, θα κόστιζε μόνο 20 δεσιμπέλ, μάλλον 20 ευρώ ένα δεσιμπέλ, 60 80 ευρώ δηλαδή συνολικά, για ένα όχημα που θα ήταν κατά 50% ε, λιγότερο ηχηρό από ό,τι τα σημερινά για τα ηλεκτροκίνητα και τα υβριδικά οχήματα ένα σύστημα θα προβλέπεται στο μέλλον. Αυτό είναι καλή συμβαστική λύση, αν και ο χρόνο θα μπορούσε να είναι συντομότερο. Και για την επισήμανση και αυτή η συμβαστική ήταν καλή, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε εντό διετία να έχει διαξαγάγει συνολική ε, μελέτη τύπου για να υποβάλει την ανάλογη νομοθετική πρόταση. Ευχαριστώ του συναδέλφου για τη συνεργασία και ελπίζω ότι θα είμαστε φιλοδοξότεροι στο μέλλον. Ευχαριστούμε κυρία Μέρκη. Ο κύριο Κάρμα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο και θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο εκπρόσωπος του συγητή και ο κ. Σταρταρέλα. Ασχολούμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό με το θέμα αυτό και δεν έχουμε απλοποιήσει τα πράγματα, ξέρετε, γιατί πρόκειται για μια ήδη προβληματική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν αρκούσαν λοιπόν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρκεί να κοιτάξουμε τον πυρήνα της νομοθεσίας αυτή στο παράρτημα και να... Φυσικά, κυρία Μερικής, μπορούμε πολλά παραπάνω να ζητάμε, αλλά πρέπει να βρούμε μια καλή ισορροπία μεταξύ χρονοδιαγράμματος και φιλοδοξίας. Πρέπει να τηρήσουμε αυτή την φιλοδοξία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επιμένει να πετύχουμε ένα σημαντικό επίπεδο μείωση στο παράρτημα. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να καταθέσουμε τροπολογίες και το πικέτ το οποίο διαπραγματευτήκαμε, θα το υποστηρίξουμε στη μορφή που έχει. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέει ο κύριος Πρόεδρος. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογίων 25 Φεβρουαρίου το μεσημέρι θα ψηφίσουμε στις 19 ή 20 Μαρτίου και προγραμματίζεται για την πρώτη ολομέλεια του Απριλίου. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα να κλείσω το σημείο αυτό της διάταξης, το 8 ε, της σημερινής διάταξης τώρα για την Διεθνή Σύμβαση του Hong Kong για τα ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση των προβλήων έχει αναβληθεί και την επόμενη συνάντηση, συνεδρίαση και η επόμενη συνεδρίαση λοιπόν θα είναι στις 6 Μαρτίου 2014. Θα έχουμε και στις 10 Μαρτίου στο Στρασβούργο α, το απόγευμα και στις 19 Μαρτίου μία συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ πολύ και πέρα στη συνεδρίαση.